If there are no Καλημέρα σα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρί τροποποίηση. Έχετε διερμηνία σε 16 γλώσσε και ω συνήθω έχετε ηλεκτρονικά διαθέσιμο το φάκελο τη συνεδρίαση ε, στο είναι εφαρμογή meeting και επίση αναμεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Επίση, έχουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων 29-30 Αυγούστου, 10 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας ε, σήμερα, θεωρείται ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις, είχαμε δύο υποεξέλιξη. Καταρχήν, ε, θέσπιση κανόνους για τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE είχε προβλεφθεί να, να λάβει χώρα αυτή τη Δευτέρα. Δυστυχώς επειδή ήταν ε, άρρωστος ο εισηγητής έπρεπε να αναβληθεί και τώρα έχει σχεδιαστεί για τις 20 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση για ε, τα πρότυπα επιδόσεων ε, για τις εκπομπές για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και τα νέα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψε με το Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου. Ο σκοπός ε, του τριμερούς διαλόγου ήταν οι δύο συνομοθέτες να παρουσιάσουν τις αντίστοιχες θέσεις τους και να δώσουν εντολή στο τεχνικό επίπεδο να εξετάσει όλες τις ε, τροποποιήσεις προκειμένου να δοθούν διευκρινήσει και να υπάρξει ευθυγράμμιση για τα τεχνικά ζητήματα. Ο δεύτερο τριμερή διάλογο ε, έχει προγραμματιστεί στο Στρασβούργο για τι 13 Νοεμβρίου. Τυχερή εγώ κατόπιν. Περνάμε στο πρώτο θέμα για συζήτηση που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Πρόκειται έκθεση του κ. Μάντλ, θέσπιση προγράμματο για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη ευρωπαϊκή στατιστική. Έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε το σχέδιο τη γνωμοδοτησής σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα για αυτή την τελευταία μέρα του Στρασβούργου. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι πρώτο στη Μέση Διάταξη, γιατί στις 9 έχω μια συνεδρίαση ε, με ε, τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κωσοκαφεδίου. Θα πρέπει να φύγω λοιπόν λίγα λεπτά πριν τις 9. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Έχω λοιπόν ένα σχέδιο γνωμοδότησης για έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάρτιση του προγράμματος, για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Αρμόδια είναι ΙΜΚΟ. Η εκεί είναι ο συνάδελφος Νικολά Νταντή. Έχουμε γνωμοδοτήσει από την Άγκρη, την ΕΚΟΝ, την Ήτρε και από εμά λοιπόν την ΕΝΒΗ. Η ΕΝΒΗ μαζί με την Άγκρη και την IMCO έχει ε, καταμεσμένη αρμοδιότητα για την τροφική αλυσίδα, τα κτηνοτροφικά μέτρα και την προστασία των φυτών. Μαζί με το πρόγραμμα του, για τις πολιτικές προοπτικές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε στις 5 Ιουνίου μια πρόταση για την εσωτερική αγορά στα πλαίσια του προγράμματος αυτού φέρονται διάφορες δραστηριότητες που μέχρι στιγμή χρηματοδοτούνταν από πέντε προηγούμενα προγράμματα και ιδιαίτερα ε, προγράμματα που αφορούν την τροφική αλυσίδα για την εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει χρηματοδότηση 4 δις εκ των οποίων 41% ε, θα πάνε για την τροφική αλυσίδα. Ιδιαίτερα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, ασθένειες και τις επιζωοτίες για να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο για τα άτομα, τα ζώα και τα φυτά και να έχουμε καλύτερη παραγωγή ε, τροφίμων. Το πρόγραμμα για την τροφική αλυσίδα αφορά και κτηνοτροφικά μέτρα για τα ζώα λοιπόν και μέτρα φυτοπροστασίας. Και αποτελείται από μονοετή ή πολιετή προγράμματα και αν έχουμε κρίσεις ή ε, απρόβλεπτα γεγονότα θα είναι δυνατόν να ληφθούν και ε, επίγοντα μέτρα. Πολύ σημαντικά από πλευράς της ΕΝΖΗ, της ΕΝΒΗ μου φαίνονται τα εξής σημεία. Για να παρατηρούμε την εφαρμογή του πολιτούς προγράμματος χρειαζόμαστε στατιστικές αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατακλειστούν οι επιχειρήσεις από γραφειοκρατία. Ένα υψηλό επίπεδο της τροφικής αλυσίδας είναι απαραίτητο για να λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά. Για παράδειγμα, ε, ε, τα φαινόμενα του φιλτρονέλη στα αυγά και το σκάνδαλο με το ε, κρέας ε, από άλογα επέδειξαν ότι οι κρίσεις και τα σκάνδαλα μπορούν να επηρεάσουν την εσωτερική αγορά και την παραγωγή. Επειδή η τροφική αλυσίδα είναι όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να ελέγχουν την τροφική αλυσίδα για να διαπιστώνουν εάν τηρούνται και επιβάλλονται τα ενωσιακά μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εισαγωγές τροφίμων. Το χρονοδιάγραμμα προτείνει ότι σήμερα στις δύο λίγη προθεσμία τροπολογιών θα ψηφίσουμε στις 6 Δεκεμβρίου, τη μέρα της ορτής του Αγίου Νικολάου. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ εκεί πρόεδρος. Ισκιώδης τώρα. Ο πρώτος είναι ο κύριος Μπάλας. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. θα επιμείνει πρώτα απ' όλα η ομάδα μου σε ένα θέμα αρχής. Δεν μπορεί να υπάρξει προστασία της υγείας των πολιτών εάν το κέρδος και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι η βασική αρχή που διέπει τις κοινωνίες μας. Το βραχυπρόθεσμο κέρδος είναι προφανώς εχθρός της υγείας των πολιτών. Δεύτερον, Μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την υγεία των πολιτών αν δεν αλλάξει ο τρόπος παραγωγής αλλά και κατανάλωσης. Αν νομίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε όπως παράγουμε και να υπάρχει τέτοια μαζική κατανάλωση χαμηλής ποιότητας προϊόντων, άλλη μια αντίφαση εις βάρος της υγείας των πολιτών. Θα πρέπει να μάθουμε να χρηματοδοτούμε τις αναγκαίες μεταβάσεις στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης προς ένα νέο πρότυπο. Ένα νέο πρότυπο που ακόμη σήμερα δεν στηρίζεται αρκετά, αρκετά θεωρούμε, από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Τρίτον, και επίσης σημαντικό, γιατί είναι κάτι που εμφανίζεται όλο και περισσότερο σήμερα και θέλω να επιμείνω, είναι οι παράνομες εισαγωγές τροφίμων και ιδιαίτερα κρέατος. Έχουμε κρέατα από την Αφρική, ζώων από τη Σαββάνα, που πολλές φορές ε, έχουν πολλά υγειονομικά προβλήματα και ποικίλα. Ιδιαίτερα το κρέας ορισμένων ε, τέτοιων ζώων ε, μπορούν να είναι φορές ασθενειών πολύ επικινδύνων. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αντιδράσουμε ταχαίως. Θα υποβάλω 14 τροπολογίες από πλευρά της ομάδας μου για να ε, ενισχύσουμε περισσότερο την προστασία των καταναλωτών. Καλύτερη εχνευσιμότητα θα ζητήσω πρώτα απ' όλα. Και έχει έχουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα με τους κώδικες που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα. Δεν είναι επαρκής. Υπάρχουν νέες διαδικασίες. Υπάρχουν τώρα οι κώδικες QR που έχουν χαμηλό κόστος και επιτρέπουν καλύτερη ανιχνευσιμότητα συμφωνούν και επιχειρήσεις από αυτού. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σήμανσης και τους ε, κωδικούς που χρησιμοποιούμε. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες και για την ε, τροφιμική αξία και για τον τρόπο παραγωγής και για τα φυτοφάρμακα. Είναι απαράδεκτο ότι στα σούπερ μάρκετ εδώ στην Ένωση δεν μας λένε τίποτα για το από πού προέρχεται, τι περιέχει αυτό το προϊόν, στην ουσία είναι αυτό προσβολή προς το καταναλωτή και κίνδυνος. Και κάτι άλλο που είναι όμως ευπρόσδεκτο. Και εγώ ασχολήθηκα ιδιαίτερα με, το, με την κατάργηση της ε, εκτροφής ζώων σε κλοβούς. Πρέπει να σταματήσει. Αυτό θα είναι καλό και για την υγιεινή, άρα και, προς την, ε, και για την υγεία μας τα ζώα τα οποία εκτρέφονται με κακό τρόπο είναι επικίνδυνα σε τελευταία ανάλυση και για τον καταναλωτή μετά την ε, διαδικασία μεταποίησης ε, των προϊόντων τους. Και δεν πρέπει φυσικά να είμαστε υπερβολικά γραφειοκρατικοί και συμφωνώ με τον εισηγητή. Πρέπει λοιπόν να εμπλακεί και η κοινωνία των πολιτών και οι ενώσει καταναλωτών. Σε πολλά κράτη-μέλη το φαινόμενο των συλλογικών προσφυγών αρχίζει και αναδύεται, το class action πρέπει και οι ενώσεις καταναλωτών και αυτές να εμπλέκονται στον ορισμό του ελέγχου των αλυσίδων παραγωγής. Δεν πρέπει να είναι μόνο το κράτος και ο κλάδος που να συνομιλούν, πρέπει να κάθεται στο τραπέζι και ο καταναλωτής. Και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Eichhout. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης και να του πω πως μπορώ να είμαι σύντομος. Θεωρούμε πως η κατεύθυνση που ακολουθεί είναι μία την οποία μπορούμε να στηρίξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Το πιο σημαντικό κομμάτι δε και στο οποίο θα θέλαμε να σταθούμε είναι πως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε πολλά σκάνδαλα με τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φιμπρονίλ, ε, το ε, κρέας αλόγου. Και αυτό δεν υποσκάπτει μόνο την εσωτερική αγορά, αλλά χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην, αγορά, στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων οι καταναλωτές και υπάρχει και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οπότε αυτά τα θέματα θα χρειαστεί να τα αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα αποδεικνύει πως έχει κανείς σκοπό να κάνει τα λόγια πράξη. Οπότε βρίσκω πολύ απογοητευτικό το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις που έκανε μειώνει τα κονδύλια για τους ελέγχους στα τρόφιμα έτσι ώστε να μην έχουμε νοθείες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θα υποβάλουμε ε, μια τροπολογία έτσι ώστε να αυξηθεί ο προπολογισμό για τα σημεία αυτά, γιατί είναι σημαντικά για να εμπιστεύονται οι καταναλωτέ στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων. Και ε, για τα υπόλοιπα στηρίζουμε ε, τον εισηγητή και στηρίζουμε και τα όσα είπε ο συνάδελφο από του σοσιαλιστέ. Οπότε πιστεύω πω για την γνωμοδότηση αυτή σύντομα θα καταλήξουμε σε μια πολύ θετική συμφωνία. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρούπαν, εκ του κύριου Πίκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου πως στηρίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ο σκοπό να στηρίξει την ε, αγορά τροφίμων. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες συνέργειες με άλλες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, τι κάνουμε με την ψηφιακή αγορά, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές εταιρείες και να προσαρμοστούν καλύτερα στην ψηφιακή επανάσταση. Εμάς μας ενδιαφέρει η προστασία της υγείας του καταναλωτή. Και όντως αληθεύει αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής. Ναι, μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, προτάσεις που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για παράδειγμα, με τις πιζωτίες ε, και το πώς έχουν εξεσπάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, να σας πω πως τα κράτη-μέλη χρειάζεται να αντιμετωπίσουν την πανόλη των χείρων, την αφρικανική πανόλη των χείρων, για παράδειγμα, και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια για την προστασία και να διατηρήσουμε τον προπολογισμό που έχουμε για την αντιμετώπιση τέτοιου ε, κρίσεων. Ε, και όχι μόνο να τον διατηρήσουμε, θα έλεγα να αυξήσουμε κιόλα, χωρί όμως με τον τρόπο αυτό παράλληλα να αυξάνουμε και το διοικητικό βάρος. Και πιστεύω πως πρέπει να τονίσουμε πως αυτό το διοικητικό βάρος δεν είναι μόνο βάρο για τι επιχειρήσει, αλλά πολύ συχνά είναι και μια επιπλέον επιβάρυνση για τη δημόσια διοίκηση. Εγώ ίσω υποβάλλω τροπολογίες αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πολλέ στον αριθμό. Any... Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιον άλλο. Εάν όχι, ο κύριος Ντιτζόλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλημέρα σας. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ξεκινήσω λέγοντας πως είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα το οποίο αντιμετωπίζει την αλυσίδα τροφίμων αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος που σχετίζεται με την εσωτερική αγορά. Αυτό αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουμε στα μέτρα που συζητάμε και κυρίως το κομμάτι το κτηνιατρικό, το κομμάτι το φυτο-υγειονομικό όπως επίσης και τους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα, που στοχεύουν στο να εξασφαλίζουμε πως οι έλεγχοι γίνονται, πως ε, είναι προληπτικοί, αλλά βέβαια πως αντιμετωπίζουμε και τις επίγουσες ε, ανάγκες που ξεσπάνε ε, με ασθένειες που εμφανίζονται, με επιδημίες, αλλά και με την εξάλληψη αυτών. Αυτή είναι η διαφορά με το επόμενο μεταξύ του επόμενου προγράμματος και του τρέχοντος και υπάρχουν και κάποια καινούρια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αλυσίδα τροφίμων. Για παράδειγμα, η ευζοία των ζώων, το θέμα των ε, τροφίμων ε, ε, που πετάμε και κάποια ακόμα τα οποία θα τοποθετήσουμε στο κείμενο. Υγεία, προστασία της ανθρώπινης υγείας και αυτό αποτελεί ένα κομμάτι των στόχων της, του προγράμματος για την ενιαία αγορά και θα προσθέσω και μια παρατήρηση για την απλούστευση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να εφαρμόσουμε κάποιες αρχές απλούστευσης στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε το πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στην προσφορά και την παράδοση αποτελεσμάτων και θα πρέπει να διευκολύνει και τη δημόσια διοίκηση έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να ε, εκτελήσουν με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Κύριος Μάντελ, για να κλείσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ επικοδομητική συζήτηση και τις πολλές ε, καλές προτάσεις. Βεβαίως ε, θα περιμένουμε ενδιαφέρον τις διάφορες τροπολογίες και χαίρομαι που κατά το μάλλον και ρητών, αλλά κατά το μάλλον θα έλεγα, πηγαίνουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Και ευχαριστώ πολύ λοιπόν και άλλη μια φορά για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών στις 2 και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, να κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Okay, so if you want to take your seats... Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε με τις ε, ψηφοφορίες. I hope you have your voting card. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες μαζί σας. Πολύ ωραία. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2020, προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μία ενιαία ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is... Λήξη. Εγκρίνεται. Το επόμενο σημείο είναι ο μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τη 15. Άρχη η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά η κάρτα μου είναι στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να λαμβάνετε υπόψη την δική μου ψήφο με την ένδειξη του εκπροσώπου των σοσιαλιστών. Τροπολογία 1. Ελέγχουμε την 1. Λήξη.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 Θα ξεκινήσουμε με την 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για να ξαναδούμε λοιπόν ηλεκτρονικά τη 13, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ την 19 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά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 εγκρίνεται. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Πάμε στην 21 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές. Τι ηλεκτρονικά παρακαλώ, την τροπολογία υπαριθμών 5. Πέρασε ψηφοφορίας εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικά παρακαλώ και την 53 τη ψηφοφορίας 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είπα 56, όχι 6. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαρθμό 7 και 58 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 8 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Υπαρθμό 8. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για να δούμε ηλεκτρονικά και την ενάτη. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 64 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 66 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική πρώτη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 ε, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, συμβιβαστική υπαριθμό 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Κύριε Λόπες, έχετε την κάρτα σας. απορρίπτεται. Παρόλο που. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Θα ψηφίσουμε και την τροπολογία 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 70. Παρακ... Α, την 69 ηλεκτρονικά. Να πούμε την 69. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας αυτής. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την τροπολογία υπάρχει 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία, συμβιβαστική υπαρθμό 5, πέρας, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ την ε, τροπολογία παριθμών 25 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 26 υπέρ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 απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπάρχουν 7 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά Άποχες. Δεν μου δείξατε τι γίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ, μάλιστα. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την τροπολογία 4. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την παρθόν 40, άρχη ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικά παρακαλώ την υπαρθμό 45. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ηλεκτρονικά για το σύνολο άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται And that concludes the... Οπότε ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες.

Um, uh, λοιπόν, ελάχιστε προποθέσει για, προϋποθέσεις για την επαναχρησιμοποίηση του ύδατο. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μπόναφε. Θα την αντικαταστήσει όμω ο κύριο Τζόφολη. Παρακαλώ, κύριε Τζόφολη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αντικαθιστώ την κυρία. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αποφύγουμε οι διάφορες απαιτήσει που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη να προκαλέσουν εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Επομένως, εγώ συγχαίρω την Επιτροπή για τη γενική παρουσίαση της πρότασης που αξιοποιεί την εμπειρία που προέρχεται από την εθνική νομοθεσία όπως από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Παρ' όλα αυτά θεωρώ απαραίτητο να παρέμβω με κάποιες τροποποιήσεις προκειμένου να καταστήσω πιο ξεκάθαρη την νομοθεσία κυρίως ό,τι αφορά τους ορισμούς για το ρόλο και την ευθύνη των διάφορων εμπλεκομένων και για τις κύριες δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου. Θεωρώ επίσης σημαντικό να διευρύνω το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού και για τις χρήσεις για περιβαλλοντικούς και αστικούς σκοπούς, έτσι ώστε να μπορούν να διευρυθούν τα ωφέλη από την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Τώρα, για να μπούμε συγκεκριμένα στις λεπτομέρειες, εφιστούμε την προσοχή στη διαφορά μεταξύ των επεξεργασμένων υδάτων ε, και ε, των υδάτων που υπόκειται σε συγκεκριμένη επεξεργασία και τα νερό από ανάκτηση που καλύπτεται από το πεδίο αυτού του κανονισμού. Συγκεκριμένα στην Ιταλική εκδοχή το να διατηρήσουμε τον ε, όρο ότι προέρχεται από επεξεργασία αντί να λέμε από ανάκτηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ερμηνεία. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να προσδιορίσουμε μεγαλύτερη ακρίβεια τους κύριους εμπλεκομένους στην διαδικασία ανάκτησης των αστικών λιμάτων. Για το λόγο αυτό μαζί με τον φορέα εκμετάλλευσης ε, ε, της ε, μονάδας επεξεργασίας, του φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης και τον τελικό χρήστη, εντάσσεται και ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής. Στο παράρτημα 2 θεώρησα απαραίτητο κατόπιν να αναφέρω με συγκεκριμένο τρόπο τους, τα ελάχιστα καθήκοντα που έχουν διάφοροι εμπλεκόμενοι. Σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσει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 συμφωνήσει με τις παραμέτρους που προτείνεται από την Κομισιόν βάσει της ε, μελέτης ε, του JRC, αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να βάλουμε και την παράμετρο σαλμονέλα για να εγγυηθούμε μεγαλύτερη διατροφική ασφάλεια για τους πολίτες, για να εκμεταλλευτούμε πλήρως ε, την δυνατότητα της ανάκτησης των αστικών λιμάτων. Είναι σημαντικό να μην περιορίσουμε την πιθανή χρήση μόνο για την άρδευση στη γεωργία, αλλά να διευρύνουμε τις χρήσεις όπως γίνεται σε διάφορα κράτη-μέλη. Όπως ε, σας είπα, για σκοπούς αστικούς παραδείγματος χάρη μπορούμε να αποτίσουμε τα γήπεδα του γκολφ ή τους πράσινους χώρους ή για περιβαλλοντικούς σκοπούς παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίσουμε την ε, αφαλάτωση κτλ δεν έχω συμπεριλάβει εναρμονισμένε παραμέτρους ε, για τι ε, βιομηχανικέ χρήσει, γιατί θεωρώ ότι τέτοια χρήση θα πρέπει να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο βάσει μεμονωμένων περιπτώσεων. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, ύπαρξη μέτρων ευαισθητοποίηση, προκειμένου να προωθήσουμε την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων που προέρχονται από την ανάκτηση των αστικών λιμάτων και ένα σύστημα που θα εγγυηθεί την υγιεινή του νερού από ανάκτηση. Επίση, δηλώνω τη λύπη μου επειδή στο πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες σε ό,τι αφορά την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα. Για τους λόγους αυτούς, εντός της ρήτρας αναθεώρησης που είναι στα πέντε χρόνια, έχω ζητήσει την δυνατότητα να προβλεφθεί νομοθετική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, έχω ζητήσει από την Κομισιόν να εξετάσει την ανάγκη ειδική ρύθμισης για την έμεση επαναχρησιμοποίηση. Αναμένω τις προτάσεις σας και είμαι σίγουρος για τη συνεργασία μας σε αυτό το σημαντικό φάκελο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Γκάμπου Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και την συγκίτρια για την εργασία που επετέλεσε, αν και δεν είναι παρούσα. Μεταξύ του 1976 και του 2006 ε, θεωρείται ότι το κόστος της ξηρασίας ανήλθε σε 100 δις ευρώ. και κυρίως ε, επηρέαζε το Νότο. Και φέτος ε, είχαμε σοβαρές ε, πυρκαγιές ακόμη και, το, και στο βορρά όπου το, η μέση θερμοκρασία είναι, ήταν 10 βαθμοί πάνω από το σύνηθε. Και πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους σε τόσο ακραίες συνθήκες. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να συμμεριστούμε την προσπάθεια αυτή με του ευρωπαίου ε, τέλου. Η κοινωνική οικονομία μα δίνει πολλέ δυνατότητε. Πρώτα απ' όλα γιατί μα επιτρέπει να έχουμε υψηλή ποιότητα στο σημείο παράδοση του επαναχρησιμοποιηθέντο ε, ύδατο. Είναι αναγκαίο λοιπόν να καθαρίσουμε του ε, συμπληρωματικού Δεν μπορεί να γίνουν όλοι οι έλεγχοι από την ε, κατάσταση επαναχρησιμοποίηση και καθαρισμού. Και γι' αυτό θα προτείνω μια σειρά τροπολογίων άλλο παράγον κινδύνου που βλέπουμε. Είναι ακριβώς ε, η ποιότητα, οι ορισμοί του επίπεδου ποιότητας. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν, αλλά να μην ε, σημαίνει αυτό ότι θα ακριβίνει τόσο πολύ το είδωρο προς επαναχρησιμοποίηση, γιατί αυτό θα αποτρέψει τους ε, χρήστες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα στόχο, γι' αυτό που είναι το 5%. Επίσης, πότε θα αρχίσει να ισχύει. η τροποποίηση, πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι ε, θα εφαρμοστούν σε χώρες που έχουν ε, μία δεκαετία μόνο χρήση ε, αυτών των δυνατοτήτων. Άρα πρέπει να υπάρξει μια δεκαετια μονο χρησης αυτων των προθεσμιών για να εφαρμοστούν τα μέτρα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και είμαστε σίγουροι ούτω ώστε ότι θα έχουμε το αναγκαίο μέσο για να έχουμε την αναγκαία ποιότητα σε επαναχρησιμοποιηθέντο ύδατο και για του ανθρώπου και για την οικονομία και έτσι να κλείσουμε τον κύκλο του ύδατο. Και ε, κάτι διαδικαστικό τώρα. Η προθεσμία για τι τροπολογίε ε, αύριο. Θέλουμε μια παράταση. Για παράδειγμα, μέχρι τη Δευτέρα. Το συζήτησα με κάποιου συναδέλφου γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε, επειδή την επόμενη εβδομάδα είναι πράσινη εβδομάδα, η Πέμπτη και η Παρασκευή λοιπόν είναι αργίε, θα μπορούσαμε λοιπόν να πάμε μέχρι τη Δευτέρα η προθεσμία, να κερδίσουμε μια εβδομάδα για να προετοιμάσουμε καλά τι τροπολογίε. Βεβαίω υφιστάμεθα πιέσει από πλευρά συνοδιαγράμματο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να εργαστούμε λίγο περισσότερο, να διαχειριστούμε καλύτερα το χρόνο μα. Η επόμενη εβδομάδα του άλλου είναι μόνο τρει μέρε. Πιστεύω λοιπόν ότι ο οργανισμός αξίζει να έχει καλές ε, τροπολογίες. Βεβαίως και οι υπηρεσίε μετάφρασης ε, έχουν τις προθεσμίες τους, αλλά και εμείς χρειαζόμαστε χρόνο για να προπαρασκευάσουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκάμπους. Ο κύριος Τόρβαλτ. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ το Γιάνν Χουίτεμα Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια για την καλή εργασία της. Υπάρχουν τέσσερα θέματα που ο κύριος Χουίτεμα θα ήθελε να τονίσει. Το πρώτο έκανε διάφορες αλλαγές στο πεδίο εφαρμογή του προτινόμενου κανονισμού. Βεβαίω να συζητήσουμε το πεδίο εφαρμογή, ανοιχτοί είμαστε. Αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσει πρακτικές ε, δυσχέρειες. Για παράδειγμα, πώς θα κατανέμεται στα γήπεδα του γκολφ το επαναχρησιμοποιηθέν Επίσης πρέπει να συζητήσουμε τη συμμόρφωση. Λέγεται ότι ο αρμόδιος της εγκατάστασης είναι αρμόδιος για, το, για την ποιότητα του ύδατος, αλλά μετά θα είναι υπεύθυνος ο τελικός χρήστης. Επίση, θέλουμε επαρκή πιλωτικά προγράμματα γιατί μπορούν ε, να δώσουν την αναγκαία όθηση για την επαναχρησιμοποίηση του χρησιμοποιηθέντο σε αστικές περιοχές ύδατο. Υπάρχουν κάποιες αλλαγέ ε, τώρα μεταξύ των, ε, των παραγόντων για την επιτήρηση και των σχέδιων για τη μετώπιση των κινδύνων μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν διάφορες διαφορές και αυτέ ε, είναι διαφορετικέ επίση από τις προτάσεις της Επιτροπής. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πιο ε, προσεκτικά αυτέ τις παραμέτρους επιτήρηση και τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων της Κομισιόν. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση της Επιτροπής ε, για την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων μας δίνει μια ευκαιρία που πρέπει να δράξει η Ευρώπη για να μειώσει την πίεση που ασκείται στους υδάτινους πόρους. Γιατί το είπαμε ότι η εξοικονόμηση του νερού μέσω της έμπαινας χρησιμοποίησης του είναι πολύ σημαντικό κυρίως ε, όταν μιλάμε για ε, αρνητικές επιδόσεις ό,τι αφορά τους υδατινούς όγκους, ε, κυρίως λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Όμως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να πράξουμε έτσι ώστε τα αστικά λίματα θα τυχάνουν της κατάλληλης επεξεργασίας και θα προσφέρουν ασφάλεια χωρίς να ρηπαίνουν τα οικοσυστήματα και τα εδάφη και χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία του πληθυσμού. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι άδειε για την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων ε, θα πρέπει να εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές μόνο αν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να σεβαστούν τα καθήκοντά τους, δηλαδή να διαχειριστούν τους κινδύνους που ενέχει η επαναχρησιμοποίηση του ρερού. Θα πρέπει λοιπόν οι φορείς εκμετάλλευσης να έχουν τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες προκειμένου ε, πλήρως να εξαλείψουν τα μικρόβια από το νερό και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει πολύ σχολαστικά να υλοποιούν τα καθήκοντα ελέγχου και παρακολούθησης και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διαδικασίες ανάντι και κατάντι της ανάκτησης των αστικών λιμάτων από στην Ιταλία Έχουμε πολύ σοβαρή ε, παραβίαση της οδηγίας των αστικών λιμάτων ε, και έχουν ξεκινήσει τέσσερις διαδικασίες επί παραβάση και ε, αφορούν πάρα πολλούς φορείς. αυτή η νομοθεσία έχει παραβιαστεί και θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή εδώ και 20 χρόνια ήδη και σε μια γενική κατάσταση από το βορρά στο νότο μας έχει οδηγήσει στο να πληρώσουμε τσουχτερά πρόστιμα. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος μας δεν θα πρέπει να είναι μόνο να δώσουμε κίνητρα για την ανάκτηση του νερού, αλλά θα πρέπει να πράξουμε έτσι ώστε να εγγυηθούμε μια συνέπεια ε, σε ό,τι αφορά το σεβασμό της νομοθεσίας ε, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλό είναι λοιπόν να δίνουμε κίνητρα προκειμένου να μειώσουμε την καταπώνηση των μάτων και προκειμένου να μειώσουμε και τον αντίκτυπο των αστικών ε, λιμάτων στους υδάτινους όγκους, όμως ε, θα πρέπει να μην υπάρχουν προβλήματα στην επεξεργασία των αστικών λιμάτων κυρίως εκεί όπου έχουμε δομικές ελλείψεις γιατί δεν είναι κατάλληλα τα συστήματα συλλογής ή γιατί δεν λειτουργούν οι εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποφύγουμε την επαναχρησιμοποίηση γιατί θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτά τα προβλήματα που είναι ανάντι της επαναχρησιμοποίησης. Το ίδιο ισχύει και εκεί όπου δεν υπάρχουν επαρκείς ικανότητες προκειμένου ε, να διαχειριστούμε τα ε, νέα απόβλητα όπως παραδείγματο το χάρη τα, ε, τα, την λιματολάσπη. Έχουμε περίπου 30 ε, εκατομμύρια τόνους ετησίως τέτοιων αποβλήτων στις πόλεις. Γι' αυτό η έγκριση για την ανάκτηση των επεξεργασμένων αστικών λιμάτων θα πρέπει να δίνεται μόνο σε τοπικό επίπεδο όταν έχουν γίνει αυστηρό σεβαστές οι διατάξεις της οδηγίας ε, για τη χρήση της ε, ε, λιματολάσπης στη Γεωργία. Και θέλω να απευθυνθώ στην Κομισιόν και να την καλέσω να υλοποιήσει την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για την λιματολάσπη, γιατί προβλέπεται να εισαχθούν κατώτετα όρια, ε, παραδείγματο χάρη για τις εγκαταστάσεις ε, και για ε, διάφορες ουσίες όπως είναι η πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακες. Σε ό,τι αφορά τώρα το σχέδιο της έκθεσης, θεωρώ ότι είναι ισορροπημένο. Σίγουρα υπάρχουν σημεία που μας βρίσκουν σύμφωνους, όπως το ότι προβλέπονται νέες υποχρεώσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής και τους τελικούς χρήστες και επίσης συμφωνούμε για την πιθανή διεύρυνση της χρήσης, όπως ε, το χάρη για αστικούς σκοπούς, ε, το να ε, ποτίζονται γήπεδα γκολ κτλ. Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε άλλα σημεία κατά την ανάλυση του φακέλου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω πως η Σολεδά Καβεσόνη, η συνάδελφος, ζήτησε να την συγχωρέσετε που δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα και να σας πω πως εμείς οι σοσιαλιστές καταλαβαίνουμε ποια είναι τα προβλήματα της πάνησης του νερού, κατάσταση που χειροτερεύει από την αλλαγή του κλίματος και που επηρεάζει όλο και περισσότερες χώρες. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση και την έκθεση Μποναφέ και συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά έχουμε και κάποια σημεία που μας ανησυχούν. Σε χώρες όπως η Ισπανία, όπου η ανακύκλωση δεν είναι χρήση, ε, δεν είναι συγγνώμη εναλλακτική λύση, αλλά είναι μια πραγματικότητα, Είμαστε το σημείο αναφοράς γιατί έχουμε το μεγαλύτερο όγκο νερού που επαναχρησιμοποιείται στην Ευρώπη, δηλαδή είμαστε περίπου στο 50% του ευρωπαϊκού συνόλου και θα πρέπει αυτή την εμπειρία τη δική μας να τη λάβετε υπόψη. Η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί είναι ουσιαστική, αλλά μας απασχολούν τα εξή. Πού θα βρίσκεται το σημείο μέτρησης, πού θα τοποθετηθεί και πού θα βρίσκεται ε, και ποια θα είναι η συνάρτησή του με το σημείο ε, έγκρισης. Επίσης, η ανάκτηση ε, των θρεπτικών στοιχείων και τέλος το διάστημα ε, που θα δώσουμε μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο κανόνας. Έχουμε και κάποια τεχνικά θέματα. Δηλαδή, το άρθρο 5, ο, ο, ο, ο και το άρθρο 6 και 7 που έχουν να κάνουν με τον φορέα του δικτύου θα πρέπει να αναλυθούν με λεπτομέρειες. Και επίσης θα πρέπει να κάνουμε τον κατάλληλο συντονισμό με την υπόλοιπη νομοθεσία που μας αφορά, δηλαδή έχουμε τον 852 του 2004 που έχει να κάνει με την υγιεινή των ε, τροφίμων. Γιατί η πρόταση όπως την έχετε καταθέσει μπορεί να μην επιτρέπει η ανακύκλωση του νερού να κάνει ε, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποκαλλιέργεια περιοχές με διαφορετικά συστήματα άρδευσης ε, έτσι ώστε στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας να μπορούμε να προσφέρουμε ε, νερό ε, στην άρδευση το οποίο έχουν προσθεθεί θρεπτικά στοιχεία. Πιστεύω ότι η επιψηλογική μελέτη επίσης δεν έχει μελετηθεί κατάλληλα και έχει υποεκτιμήσει το κόστος και να μιλήσω για το θέμα της επαναχρησιμοποίησης νερού για να καλύψουμε ε, το θέμα της ε, λειψιδρίας και να δούμε πώς επηρεάζονται από αυτήν ο βιομηχανικός και ο γεωργικός κόσμος. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πως χρειάζεται να έχουμε ψηλά επίπεδα προστασίας για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, παράλληλα όμως τονίζοντας πως η πρόταση θα πρέπει να λάβει υπόψη την εμπειρία και την εφαρμογή στην πράξη από τις χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει πιο πολύ στο θέμα αυτό, όπως είναι η δική μας περίπτωση ε, τη στιγμή που προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα θέματα στην Ελλάδα. στην Ευρώπη. Επομένω, πρέπει επίση να έχουμε κατάλληλο χρόνο για τη θέση σε ισχύ και αυτό ο κανονισμό ε, πρέπει να εφαρμοστεί με σωστό τρόπο. Σα ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Λίζα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την εισηγήτρια, παρά το ότι αποσιάζει. Μία ερώτηση μόνο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανονισμό. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, για τη χρήση του ύδατος ε, στην ε, Ευρώπη. Γιατί να μην επιλέξει άλλο νομικό μέσο για να είναι μεγαλύτερη η ευελιξία. Και επίσης, ο Φραντσές Καμπούς είπε κάτι. Εμείς, ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, θέλουμε να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Για μας είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση όμως. Αυτή τη βδομάδα ε, είχαμε 6-7 θέματα στην Ολομέλεια και την έκθεση downtown λοιπόν για το νερό. Και τώρα μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε τροπολογήσει για αυτό το θέμα. Στηρίζω αυτό που είπε ο κύριος ε, Γκαμπούς να μας δώσετε κάποιες μέρες παραπάνω για τις τροπολογίες. Εντάξει, υπάρχει ένα μικρό κίνδυνος, δεν μην να το βάλουμε στην ε, ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, αλλά νομίζω ότι αν μετά επιταχύνουμε θα προλάβουμε παρόλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να σας πω πως το θέμα αυτό της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων είναι κάτι που ανησυχεί πολλούς ε, τις ε, αρχές ε, υπεύθυνε για το νερό, τους ε, γεωργούς, τη δημόσια διοίκηση. Ξέρετε πως υπάρχει θέμα και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε χρηστή διαχείριση των υδάτων και θα πρέπει παρόλα αυτά να έχουν για την άρδευση καλή ποιότητα νερό οι γεωργοί και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για θέματα υγείας του Ευρωπαίου καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λογική ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ποιότητας των ευρωπαϊκών τροφίμων και της ανάγκης να έχουμε μια πολιτική που θα δώσει κίνητρα ε, στους γεωργούς να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο νερό αντί ε, νερό από τη βρύση. Θα ήθελα η συγγετρία να προσέξει ε, τον ορισμό των ευθυνών ε, καθενός από τους παίκτες και των εμπλεκόμενων ε, σε αυτή τη διαδικασία. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναλάβουν την αξιολόγηση κινδύνου και να αξιολογούν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιάσει αυτό το νερό που επαναχρησιμοποιείται. Επίσης, η αποθεματοποίηση και αποθήκευση αυτού του νερού, γιατί πολλές φορές το ανακυκλωμένο το νερό το χρησιμοποιούν οι γεωργοί αμέσως, άλλες φορές όμως το αποθηκεύουν σε δεξαμενές. Ξέρετε πως αυτό μπορεί να έχει κάποιες ποιοτικέ επιπτώσεις, να χειροτερεύει η ποιότητα τη στιγμή της ε, αποθήκευσης. Και πολλές φορές ε, δεν συζητάμε για το θέμα του κόστους όταν μιλάμε για μια πολιτική με κίνητρα. Θα πρέπει λοιπόν η ποιότητα ε, να λάβει υπόψη τον πραγματικό κίνδυνο, τον υγειονομικό και να δούμε και πώς αυτό θα επηρεάσει το κόστος. Στις 8 το μηνός εμείς ε, ε, κάναμε μια συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους και φαίνεται ξεκάθαρα πως θα πρέπει να συνεχίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζουμε την έρευνα στο θέμα αυτό και, φανταζ... και έχω κατά νου κυρίως εδώ το πρόγραμμα Horizon 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Είμαι επικεφαλής της μονάδας για το νερό στην ε, DGNV και μία από τις συντάκτρες αυτής της πρότασης, οπότε είμαι πολύ ε, ικανοποιημένη που, είμαστε, που είμαι εδώ σήμερα και ευχαριστώ όλα τα μέλη που στήριξαν τις προτάσεις μας. Ε, την έχουμε προετοιμάσει σε πολύ βάθος, ήταν χρόνια στα σκαριά και την επιδοσιολογική μελέτη την πήραμε πέρυσι το καλοκαίρι και ήταν ένα καλοκαίρι ε, μεγάλης ξηρασίας στην Ευρώπη, κάτι το οποίο έχουμε κατά νου, γιατί ε, την Άνοιξη φέτος, όταν παρουσιάσαμε την ε, πρότασή μας, είχαμε πει τι θα γίνει το καλοκαίρι το 2018. Και το 2018 για πολλές χώρες στην Ευρώπη ήταν πολύ διαφορετικό, όχι μόνο στον Νότο. Θα, ξέρετε και εσείς πως στο παρελθόν τη χρήση, την επανάχρηση νερού την είχε κάνει κυρίως οι χώρες του Νότου. Αλλά πρέπει να σας πω πως οι χώρες όπως η Σουηδία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Εστονία, Δανία, είχαμε τεράστιο θέμα. Οπότε πιστεύουμε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναλάβουμε δράση. Η πρόταση αυτή είναι στο τραπέζι για περαιτέρω συζήτηση, γιατί θέλουμε να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί το θέμα της λεψιδρίας. Η πρόταση αυτή είναι ένα μικρό βήμα, όμως είναι το πρώτο βήμα. Είναι ένα ξεκίνημα και μπορεί να μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είδατε την έκθεση της IPPC για την αλλαγή του κλίματος αρχές Οκτωβρίου και η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση υδάτων ήδη για να μην έχουμε περισσότερες βλάβες στο μέλλον. Η πρότασή μας αναγνωρίζει πως δεν επιθυμούν όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν σε επαναχρησιμοποίηση του νερού. Και αυτό απαντά στην ερώτηση Λίζε. Για το λόγο αυτό είπαμε πως μπορούμε να έχουμε κανονισμό και όχι οδηγία, γιατί στον κανονισμό έχουμε άμεση εφαρμογή και όπου χρειαστεί θα εφαρμόζεται. Όπου υπάρχει επιθυμία να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή το βάρος της μεταγραφής στο Εθνικό Δίκαιο για τα κράτη-μέλη. Άρα δεν έχουμε αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και το κόστος που προκύπτουν από μια τέτοια διαδικασία. Και με τον τρόπο αυτό ε, θα γίνουμε ε, ε, πιο γρήγοροι ε, και δεν θα επιβάλλουμε και κάτι σε όσους δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν την πρόταση. Είναι ε, μία πρόταση που στοχεύει κυρίως στην αγρο... γεωργική άρδευση. Γιατί? Γιατί εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η παρέμβασή της δικαιολογούνται λόγω της διάστασης εσωτερικής αγοράς, το οποίο το πολύ σήμερα, και έχουμε προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα άρδευσης με τέτοιου είδους ύδατα που κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. Οπότε, ναι, έχουμε ευρωπαϊκή ε, διάσταση. Δεν έχουμε κάνει επιπτωσιολογική μελέτη σε άλλους κλάδους που αναφέρθηκαν σήμερα. Για παράδειγμα, η άρδευση των γηπέδων γκολφ, ε, πάρκα ε, κτλ. Αλλά θεωρούμε πως αποτελεί εξαιρετική πρακτική. Κάπου γίνεται, αλλά δεν έχει την ίδια ευρωπαϊκή διάσταση που έχει η άρδευση στη γεωργία. Άρα λοιπόν εκεί δεν είναι εύκολο να ζητήσουμε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει. Αντίθετα, εμείς θέλουμε με κάθε τρόπο να προωθήσουμε το θέμα αυτό και στην, στο σχέδιο δράση για την κυκλική οικονομία εμείς έχουμε στρατευθεί ε, σε μια ευρεία προσέγγιση του θέματος της χρήσης των υδάτων. Ένα στοιχείο είναι η σημερινή πρόταση, αλλά έχουμε πολλά ακόμα όπως είπε και ο κύριος Ντάντα, έχουμε και τις επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία. Πιστεύουμε πως η πρότασή μας έχει το δυναμικό να βοηθήσει την Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά και σε παγκόσμιο επίπεδο να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Να γίνουμε παγκόσμιος παίκτη σε αυτή την τεχνολογία. Η πρόταση, καταρχήν, θέλει να βοηθήσει το περιβάλλον είδατε τα νούμερα, είδατε τι μπορεί να γίνει και ξέρετε ποια θα μπορούσαν να είναι τα αποτελέσματα. Θα έχουμε λιγότερες διαρροές και ε, πιο αποδοτική χρήση, προσφέροντας και μία βιώσιμη ε, ποσότητα νερού για άρδευση στη γεωργία. Άρα λοιπόν θα μπορούν οι γεωργοί να λαμβάνουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και η διαχείριση ε, του διαθέσιμου ε, νερού να γίνεται πιο αποτελεσματικά από αυτούς. Εμείς δεν ρυθμίζουμε τίποτα παραπάνω από αυτούς που παράγουν αυτό το επαναχρησιμοποιούμενο νερό. Καλύπτουμε δηλαδή ένα νομικό κενό το οποίο είναι η κάλυψη ε, του ε, νερού που προκύπτει από τις οδηγίες για τα υγρά απόβλητα το οποίο σέβεται τις προδιαγραφές για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και παράλληλα έχουμε και την νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων, η οποία όπως είπατε και εσείς θα ρυθμίζει ποιοι είναι οι τελικοί καταναλωτές αυτών των προϊόντων από ανακυκλωμένο ε, νερό άρδευσης και τι μπορεί να κάνουν οι γεωργοί και πώς θα γίνεται και η κατανομή αυτού του νερού. Άρα λοιπόν μόνο ε, φορεί διαχείριση στα κράτη-μέλη, τελειώνει δηλαδή στο σημείο συμμόρφωση, για να το πω διαφορετικό, το οποίο είναι ε, το σημείο διάθεση τη μονάδα ανακύκλωση. Τώρα, για τους γεωργούς και το κατά πόσο μπορούν να έχουν διαφορετικές πηγές ε, για νερό άρδευση. ναι, εμείς δεν τους περιορίζουμε καθόλου με την πρότασή μας. Το μόνο που λέει η πρόταση είναι, αν χρησιμοποιεί κανεί ανακυκλωμένο νερό από αστικά απόβλητα, θα πρέπει να σέβεται μια σειρά από προδιαγραφές και ναι, μπορεί να απολύεται προς αυτό το στόχο. Ο Γιωργός, αν αποφασίσει να το αναμίξει με άλλες πηγές υδάτων, δηλαδή μπορεί να έχει συλλέξει νερό από κάπου, αυτό ρυθμίζεται από τον κανονισμό ε, για την ασφάλεια των τροφίμων, όπου υπάρχουν σχετικές διατάξεις για το καθαρό νερό που πρέπει να χρησιμοποιείται για την άρδευση. Οπότε δεν μπορούμε να ε, νομοθετούμε δύο φορές ε, και για το λόγο αυτό περιοριστήκαμε. για τις προθεσμίες που αναφέρθηκαν. Βεβαίως είναι απαραίτητο να δώσουμε χρόνο σε όσους είτε θέλουν να, να ξεκινήσουμε μια νέα επιχείρηση ή για όσους έχουν επιχείρηση αλλά θέλουν να την αναβαθμίσουν για να παράγουν άλλες ποιότητας νερό. Αυτό θα αποφασιστεί και είναι κομμάτι της διαδικασίας συναπόφασης. Πρέπει όμως να θυμόμαστε πως μετά ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να τρέξει και μετά θα τον αξιολογήσουμε και θα κάνουμε αλλαγές. Οπότε αυτό θυμηθείτε το όταν θα αποφασίσετε πόσο χρόνο θα δώσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και μία αναθεώρηση αφού τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τζοφόλη, θέλετε να επανέλθετε. Όλοι γνωρίζετε τη συνάδελφο Μποναφέ, επομένω είμαι σίγουρο ότι θα συμπεριλάβουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι παρατηρήσει σα και θα φτάσει σε μια σύνθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα το αίτημα παράταση χρόνου για την κατάθεση τροπολογιών, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι λογική η πρόταση αυτή. Δεν ξέρω ποιο ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα και αν είναι συμβατό με τη βούληση να το συζητήσουμε και στην Ολομέλεια εγκαίρω. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το αίτημα που κατατέθηκε, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 5η Νοεμβρίου στις 11 και θα ψηφίσουμε στην ΕΝΒΗ 21-22 Ιανουαρίου. Διαφορετικά δεν είναι σίγουρο ότι θα προλάβουμε την Ολομέλεια του Φεβρουάριου λαχθάιν αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσέλευσή σας. Θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρίασή μας.